Ο τρίτος στόλος φτάνει στη Γάζα. Και θα ήθελα να σας καλέσω όλους να στηρίξετε αυτή την ειρηνική εκδήλωση για να δείξουμε στους πιο φτωχούς της Γάζας ότι δεν τους έχει ξεχάσει η διεθνής κοινότητα και ότι κρατάμε τις αποστάσεις μας απέναντι στις απειλές του Ισραήλ που λέει ότι θα περάσει σε νέες δράσεις όπως το έκανε και πριν από πέντε χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί σκοτώθηκαν. Θέλω να απευθυνθώ εδώ στο Συμβούλιο πρέπει ειλικρινά να βρούμε λύσεις προκειμένου να υπάρξει ευκαιρία να αλλάξει η κατάσταση εκεί. Σας ενημερώνω ότι στις 15 Ιουνίου 2015 ε, δημιουργήθηκε μια νέα πολιτική ομάδα, η Ομάδα Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, (ENF) ε αποτελείται από 36 βουλευτές. Η δήλωση σύστασης αυτής της πολιτικής ομάδας προβλέπεται από τον κανονισμό και μου διαβιβάστη. Οι αρμόδιες αρχές